Ε. Το επόμενο σημείο της μερίσιας διάταξης είναι κοινή συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε μία δήλωση της εκπροσώπου της Αντιπροέδρου της Επιτροπής σε σχέση με την ετήσια έκθεση για τα δικαιώματα του ανθρώπου για το έτος 2008 και την έκθεση της κυρίας Χάουταλα για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς επίσης και κάποιες προφορικές ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή για το εμπόριο εργαλείων βασανιστήριων. Επομένως, πρώτα απ' όλα θα ακούσουμε την παρέμβαση της συναδέλφου Χάουταλα για τέσσερα λεπτά από την ιδιότητά της ως εισηγήτριας. Πρέπει να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για τη συζήτηση αυτή που μας ε, Τρέπει να συζητήσουμε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εδώ είναι η κυρία Άστον, είπατε εκπρόσωπος, η οποία θα παρουσιάσει την ετήσια έκθεση. Αλλά θα ήθελα να παρουσιάσω την έκθεση μου, του οποίου ο στόχος είναι να βελτιώσουμε την θέση των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ξέρετε ότι μας απευθύνονται αιτήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από διάφορες πλευρές και εδώ μιλάμε για άτομα που διακινδυνεύουν τη ζωή τους προσπαθώντας να προασπίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπως σας είπα προέρχεται αυτό από όλες τις ε, υπήρους και πολλές φορές είναι δύσκολο να διευκρινίσουμε τι είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Είναι δύσκολο να το διευκρινίσουμε, αλλά μιλάμε εδώ για άντρες και γυναίκες οι οποίοι αποποιούνται την σωματική τους ακαιρεότητα για να προσπίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχω την τιμή να καταρτήσω αυτή την έκθεση γιατί μιλάμε εδώ για την προάσπιση των δικαιωμάτων τα οποία είναι ε, ε, κατά ή στην, το επίκεντρο της πολιτικής μας. Πρέπει όμως να κάνουμε πολύ περισσότερο. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπάρχει η κυρία Άστον, η ύπατη εκπρόσωπος και πρέπει να συνεργαστούμε πολύ πιο στενά. Θα πρέπει επίσης να πρασιάσουμε ε, τις ενέργειες για να μπορέσουμε να συσφίξουμε τις ε, σχέσεις μας με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις διάφορες οργανώσεις. Συγχρόνως υπάρχει μία νέα κατάσταση με την ε, ψήφιση της συνθήκης της Λισαβόνας και πρέπει να μπορούμε να υποφεληθούμε κατά τρόπον ώστε τα ανθρώπινα δικαιώματα να τη χάνουν προασπίσεως από όλες τις πλευρές του κόσμου. Υπάρχει μια σειρά ιδεών που απαριθμίζονται. Ξέρω ότι δεν είναι όλες νέες, αλλά πιστεύω ότι όλα αυτά τα έχουμε ε, σκεφτεί πάρα πολύ προσεκτικά και το βασικό είναι να το εφαρμόσουμε διότι ε, ε, ήδη υπό την Τσεχική Προεδρία είχαμε συζητήσει τη δημιουργία ενός δικτύου ε, πόλεων καταφυγίου. Δηλαδή όταν υπάρχει ένας προσπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ο οποίος κινδυνεύει πραγματικά να μπορεί να στραφεί προς το δίκτυο αυτό. Και θυμάμαι ε, τι απήχηση είχαν όλα αυτά στις οργανώσεις. Πρέπει όμως ίσως να εντείνουμε τις προσπάθειές μας περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Επίσης αναφερόμαστε στους προσπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βλέπουμε ότι αυτοί οι προσπιστές πρέπει να μπορούν να εγκαταλείψουν τη χώρα στην οποία διαβιούν και εδώ ίσως οι Υπουργοί Εξωτερικών Υποθέσεων θα πρέπει να συνεργαστούν στενά με τους Υπουργούς Εσωτερικού ιδίως όσον αφορά τις αποφάσεις για τις θεωρήσεις κατά τρόπον ώστε να υπάρξει μία ε, επιτάχυνση της διαδικασίας. Στο σχέδιο αυτό εκθέσεως επανερχόμαστε στις εξωτερικές δράσεις στο κοινοβούλιο στις εξωτερικές εκπροσωπήσεις, δηλαδή σε όλα αυτά τα οποία ουσιαστικά ευθύνονται για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και επιμένουμε ε, επίσης ε, ε, για το ότι ο ύπατος εκπρόσωπος όταν μετακινείται πρέπει να συναντά τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ε, όλους αυτούς οι οποίες έχουν σχέσεις με ε, τα ε, δικαιώματα του ανθρώπου. Τώρα έχει το λόγο ο κύριος Αλμπερτίνη ως συντάκτης μίας εκ των προφορικών ερωτήσεων. Έχει στη διάθεση του 5 λεπτά. Πρόεδρε, το άρθρο 5 της ε, Διεθνούς Δήλωσης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων λέει ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να υποστεί βασανιστήρια, ε, τιμωρία, βία, και απάνθρωποι. Αυτό ισχύει για οποιαδήποτε ε, περίσταση ως διεθνές δίκαιο και άρα ισχύει για όλα τα κράτη, όχι μόνο η Διεθνής Δήλωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αλλά και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση ε, υποστηρίζουν την ίδια προστασία του ανθρώπου κατά των βασανιστήριων. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, λαμβάνει σοβαρά υπόψη τι υποχρεώσει τη αυτέ. και μάλιστα στην εορτασμό της ημέρας ανεβάσανιστήριων την επόμενη εβδομάδα θεωρούμε πως αυτό θα πρέπει να ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ακριβώ για να σεβαστούμε αυτέ τι νομικέ και ηθικές υποχρεώσει. χρειάζεται προσεκτικός έλεγχο το υλικό που στόχο έχει τα βασανιστήρια. Ο κανονισμός αποτέλεσε ένα μεγάλο βήμα μπροστά, όπως επιβεβαίωσε και ο ειδικό εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση των βασανιστήριων. Αποτελεί πρότυπο όσον αφορά τη διεθνή νομοθεσία για τα θέματα αυτά. Δυστυχώς η εφαρμογή αυτού του κανονισμού δεν ήταν υποδειγματική όπως ήταν η υιοθέτησή του. Μόνο επτα κράτη-μέλη έχουν ε, παρουσιάσει μία από ή περισσότερες από τις, διεθν... Ε, τις αιτήσεις εκθέσεις που, που, που περιλαμβάνονται, προβλέπονται μάλλον από τον κανονισμό και προβλέπουν τον έλεγχο εισαγωγής ή εξαγωγής ε, εργαλείων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για, τα, για βασανιστήρια. Τέτοια αξιολόγηση θεωρείται απαραίτητη για να αξιολογηθεί πλήρη σεβασμός αυτού του κανονισμού. Από την ανάλυση προκύπτουν διάφορα αιτήματα όσον αφορά την τελική χρήση και τον προορισμό των, ε, εμπορευμάτων. Οι αρχές που είναι αρμόδιες για τις εξαγωγές θα πρέπει να προβαίνουν σε πολιτική αξιολόγηση εις βάθος πριν να προχωρήσουν. Τα κράτη-μέλη τα οποία επίσης έχουν διακοινώσει τις πληροφορίες σε σχέση με τις κυρώσεις που θα πρέπει να εφαρμοστούν για την παραβίαση των διατάξεων του κανονισμού του Συμβουλίου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 16 του ίδιου κανονισμού, δεν είναι πολλά. Ε, πέντε χρόνια μετά από την εφαρμογή του κανονισμού, κατάλογος των εμπορευμάτων που έχουν εντοπιστεί ε, στον κανονισμό πρέπει να ενημερωθεί και ο άνθρωπος πάντοτε μπορεί να είναι πολύ βίος και φαίνεται πως ε, η ανθρώπινη φαντασία στο πώς να επιφέρει ε, πόνο στον άλλο, στο συνάνθρωπο είναι ατελείωτη. Θα πρέπει λοιπόν να συμβαδίσουμε με τις τεχνολογικές εξελίξεις σε αυτό το θλιβερό πλαίσιο. Γι' αυτό θα πρέπει και να θυγεί και το θέμα μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ζητήσουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να δείξουν ότι θα είναι στο ύψος των περιστάσεων. Ως Ευρωβουλευτές, καθήκον μας είναι να εξασφαλίσουμε την σωστή υπεύθυνη λειτουργία των θεσμών και γι' αυτό και θέλουμε λεπτομερείς πληροφορίες για το τι έχει γίνει μέχρι στιγμής ώστε να γίνει πλήρως σεβαστός και να τηρηθεί ο κανονισμός αλλά και όσον αφορά τα μέτρα που επιτρέπουν τη βελτίωση της κατάστασης στο μέλλον. Δεχόμαστε ευνοϊκά σε πρώτο βήμα την απόφαση της Επιτροπής που εποπτεύει την εφαρμογή του κανονισμού στο τέλος αυτής της, ε, του μήνα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κανονισμός 1236 ε, του 2006 του Κοσυμβουλίου να μην αντιπροσωπεύει μόνο ωραία λόγια, αλλά ένα θεμελιώδες μέσο το οποίο θα πρέπει πλήρως να εφαρμοστεί και αμέσως. Σας ευχαριστούμε κύριε Αλμπερτίνη. Το λόγο συντάκτη ε, μια άλλη προφορική ερώτηση έχει το λόγο ο συνάδελφο Μορέιρα για πέντε λεπτά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Αντιπρόεδρε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είπατε εκπρόσωπε τη Ένωση για τι Διεθνεί ε, Σχέσει, ε, κυρίε και κύριοι βουλευτές. Ε, εγώ, εξ ονόματο της Επιτροπής Διεθνού Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θέλω να αιτιολογήσω με κοινή προφορική ερώτηση όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού που απαγορεύει ή ορίζει το διεθνέ εμπόριο προϊόντων ή εργαλείων που στόχο έχουν ή που μπορεί και να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή της ε, ε, θανατικής ποινής, βασανιστήριων ή άλλων ε, απάνθρωπων ε, πρακτικών. έχουν εκφραστεί ανησυχίε από κυβερνήσει και από ΜΚΟ, ιδιαίτερα για την χρήση αστυνομικών εξοπλισμών και εξοπλισμών ασφαλείας για ενέργειε για βασανιστήρια. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, θέλει να ζητήσει από την Κομισιόν μία πρόταση για ευρωπαϊκή νομοθεσία που ρυθμίζει το εμπόριο τέτοιων ε, εργαλείων. Η Κομισιόν το 2005, μάλλον το επόμενο έτος, μας ε, πρότεινε τέτοιο κανονισμό και εγκρίθηκε το 1236 το 2005 ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, επιβάλλεται δεσμευτικό έλεγχο για μια ολόκληρη σειρά εξοπλισμών που, μπορούν να χρησιμοποιη... που συχνά μάλλον χρησιμοποιούνται και παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά που δεν αναφέρονται στου καταλόγου του στρατιωτικού εξοπλισμού, ούτε ε, περιλαμβάνονται στι στρατηγικέ εξαγωγέ των κρατών μελών. Άρα λοιπόν απαγορεύεται η εξαγωγή και η εισαγωγή προϊόντων που στόχο έχουν τον, αυτή τη χρήση και ζητά έγκριση για την εισαγωγή-εξαγωγή προϊόντων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τέτοιους στόχους. Άρα λοιπόν χρειάζεται η έγκριση των κρατών μελών και η υποπτία για την εφαρμογή αυτών των κανόνων. Φαίνεται πως το 2010 έχει γίνει μια πολύ σημαντική πρόοδος όσον αφορά την προστασία Τη προσωπική ταυτότητας, της εκαιρεότητας και της ανθρώπινης ζωής και που συμπεριλαμβάνονται και στο Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αλλά και στην Διεθνή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και στο Συμβούλιο τη Ευρώπη. Αυτό ο κανονισμό χειροκροτήθηκε από ειδικού και από ειδικού ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όπω ήδη αναφέρθηκε και ο ειδικό ε, εισηγητή του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια θεωρεί πως αυτό το, αυτός ο κανονισμός μπορεί να χρησιμεύσει ως πρότυπο ε, παρόμοιες για χώρες άλλων περιοχών. Όμως, τι ισχύει, τι, μάλλον τι ωφελεί ένας τέτοιος κανονισμός αν δεν εφαρμόζεται ε, σωστά. Τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή του, αλλά δεν υποβάλλουν τις εκθέσεις που πρέπει όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού. Είναι πραγματικά αυτό απογοητευτικό. Το να γνωρίζουμε ότι μόνο 7 χώρες έδωσαν πληροφορίες για τις αποφάσεις που έλαβαν σε σχέση με τους συγκεκριμένα άρθρα. Και δεν έχουμε παρά μόνο δύο εκθέσεις ε, και με ελλειπείς πληροφορίες όσον αφορά την ε, κατάσταση αυτή. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δεχόμαστε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιτρέπουν να κλείνουν τα μάτια στην κατασκευή και στο διεθνές εμπόριο των προϊόντων που απαγορεύονται ή, εν πάση περιπτώσει, διέπονται από αυτό το κανονισμό. Καταρχήν, τα κρατημέλη θα πρέπει ρητά να είναι κράτη τα οποία πληρούν τις υποχρεώσεις τους όπως προβλέπονται από τον κανονισμό και θα πρέπει εγκαίρως να υποβάλουν ε, αιτήσεις εκθέσεις όσον αφορά τις δραστηριότητε αυτές και να δίνουν πληροφορίες που να επιτρέπουν το δημόσιο έλεγχο όπως δει, συμπεριλαμβάνοντας αυτές τις εκθέσεις ως μήνυμο τον αριθμό των εισαγωγών ή των εισαγωγών τα, στοιχεία, τα χώρες προέλευσης και, και προορισμού για όλα αυτά τα εργαλεία. Η έκθεση θα πρέπει να αναφέρει όλες αυτές τις δραστηριότητες και θα πρέπει να γνωρίζουμε επίσης ποια μέτρα έχουν ληφθεί ή προβλέπονται για τις περιπτώσεις παραβίασης του κανονισμού. Τέλος, υπάρχουν προβλέψεις για ενημέρωση και για να εισαχθούν εδώ περισσότερες ε, ρυθμίσεις στα παραρτήματα και για να ανανεωθούν τα παραρτήματα αυτά. Κυρίες και κύριοι, αυτός ο κανονισμός είναι απόδειξη ότι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να απαιτήσει την απαγόρευση ε, ε, εμπορίου τέτοιων εργαλείων. Δεν μπορεί να επιτρέπεται το εμπόριο μέσων ε, θανάτωσης ή βασανιστήριων. Θα πρέπει σοβαρά να εφαρμοστεί αυτός ο κανονισμός ώστε να χρησιμεύσει ως πρότυπο όπως θέλαμε στην Ένωση, αλλά και για χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στην κυρία Άστον για να κάνει τη δική τη εισαγωγή και να απαντήσει στα όσα ακούστηκαν. Κυρία Άστον, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ, χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίνετε η δυνατότητα να συζητήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολλέ φορέ έχει δηλώσει τη δέσμευσή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό και συμμερίζομαι πλήρω ε, ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι στο επίκεντρο της ταυτότητάς μας και των ε, όσων κάνουμε εδώ, σε διεθνές επίπεδο το κράτος δικαίου, η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τα 27 κράτη-μέλη είναι μια, ε, είναι μια ιστορία επιτυχίας και είναι και πηγή έμπνευση ε, για πολλούς άλλους. Επομένως είναι λογικό να θέλουμε να έχουμε μια ισχυρή δέσμη μηχανισμών ε, για να προαγάγουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, τους τελευταίους 18 μήνες έχουμε παράσχει 235 εκατομμύρια ευρώ ε, για 900 σχέδια από μη κυβερνητικέ οργανώσεις σε 100 χώρες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικός project και πρέπει να συνεχιστεί. Δεν είμαστε όμως ο μόνος παράγοντας ε, και δεν είναι και η μόνη ε, επιτυχημένη ιστορία αυτή η δική μας. Θα πρέπει λοιπόν να διερωτηθούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Είναι μεν οικουμενικά τα δικαιώματα του ανθρώπου, αλλά δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε μια μονομερή προσέγγιση. Σίγουρα δεν θα πρέπει να αλλάξουμε το μήνυμα για τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά θα πρέπει να είμαστε πιο ευφυεί ε, στην εκπομπή του μηνύματο αυτού και θα πρέπει να κάνουμε πρόοδο. Θέλουμε την ατζέντα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να την αντιμετωπίσουμε εστιασμένα αποτελεσματικά. Θα πρέπει να στοχεύσουμε τι προσπάθειέ μα ε, με βάση την κατανόηση τη χώρα που έχουμε κάθε φορά ε, απέναντί μα και να επικεντρωθούμε επίση στα αποτελέσματα. Τα προηγούμενα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν ζητήσει για περισσότερη πληροφόρηση και καλύτερη εκτίμηση τη αποτελεσματικότητα των πολιτικών μα. Συμφωνώ και συμμερίζομαι τι ανησυχίε σα. Πρέπει να κρίνουμε τι προσπάθειέ μα μέσω των αποτελεσμάτων του ακόμη και αν πρόκειται για μια επένδυση μακροπρόθεσμη το έργο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το έργο της Προέδρου ε, της κυρίας Χάουταλα, δηλαδή η έκθεσή της για τους των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα των προσπαθειών. Χαιρετίζω την έκθεση και τα πορίσματά της και ευχαριστώ όλους όσους ε, συνέδραμα στις προσπάθειες για τη σύνταξη της έκθεσης. Πρέπει να καταστήσω σαφές ότι θα συνεχίσω να συναντώ παράγοντε ε, τη κοινωνία των πολιτών, υπερασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στι Βρυξέλλε και στο εξωτερικό. Το έχω πράξει ήδη στη Γάζα, στην Κίνα και πιο πρόσφατα στι Βρυξέλλε. Αναμένω επίση και του συναδέλφου μου από τι αντιπροσωπείε στι Βρυξέλλε και εδώ να πράξουν το ίδιο. Ένα καλό παράδειγμα του να είμαστε ευφύ και καλά οργανωμένοι είναι το έργο μα για την πρόθεση τη επικύρωση ε, του καταστατικού τη Ρώμη ε, εν ώψη τη συνδιάσκεψη Χαμπάλ. Θέλουμε λοιπόν να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη και με την Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σα δώσω και ένα επιτυχημένο παράδειγμα. Όταν επισκέφθηκα τον προηγούμενο μήνα τη Χέλη, ε, συζήτησα διάφορα ζητήματα ε, στα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε ενισχυμένη ε, συνεργασία. Και ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, ίσως προτεραιότητα, ήταν το θέμα της πειρατείας. Ε, ο κύριος Μισελ ε, κλήθη να υποβάλει το υπόμνημα αυτό στις, στο Κοινοβούλιο και έχω λάβει επίσης και επιβεβαίωση έγγραφη από την κυβέρνηση της χώρας αυτής ότι έχει ξεκινήσει τη σχετική διαδικασία. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα για την κατάργηση της θανατικής ποινής σε παγκόσμιο επίπεδο. Θέλω να σας πω ότι για μένα είναι και προσωπική προτεραιότητα η κατάργηση τη θανατική ποινή. Θα φροντίσω λοιπόν να γίνουν ε, πρόοδοι και σε διμερέ και σε πολυμερέ επίπεδο και σε ε, τέτοια βήματα συζήτηση. Το Σεπτέμβριο θα γίνει το πρώτο βήμα. Ε, γνωρίζετε ότι θέλουμε να έχουμε μια πιο συνεκτική, μια πιο αποτελεσματική εξωτερική πολιτική στο πλαίσιο ε, και της διαδικασίας Λισαβόνας. Ε, θέλουμε λοιπόν να προαγάγουμε τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Και αυτό θα διατρέχει όλες μας τι πολιτικές, οτιδήποτε κάνουμε σε εξωτερικό επίπεδο η Υπηρεσία για τι εξωτερικέ δράσει ε, όταν πλέον συσταθεί και λειτουργήσει, θα μα δώσει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε το δυναμικό μα, να μιλήσουμε με μία φωνή. Και στο πλαίσιο αυτής της ε, ολοκληρωμένης δομή, η υπηρεσία θα φροντίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα να αποτελούν ε, μία διάσταση σε όλε μα τι πολιτικέ και στην ΕΠΑ και στην ανάπτυξη και στο εμπόριο. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ και στην προφορική ερώτηση τώρα σε αυτό το πλαίσιο, σε ό,τι αφορά το εμπόριο εργαλείων βασανιστήριων. Είμαστε δεσμευμένοι για την καταπολέμηση των βασανιστήριων σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Οποιαδήποτε έλλειψη ή ανεπάρκεια για την εφαρμογή του κανονισμού 1236 του 2005 πραγματικά πρέπει και θα αντιμετωπιστεί. Και σε αυτό το πνεύμα καλέσαμε, την, καλέσαμε τη Διεθνή Αμνηστία μεταξύ άλλων να παρουσιάσει τα απορίσματά της ε, στη Ρυθμιστική Επιτροπή με τα κράτη-μέλη. Και σε αυτό το τομέα και σε άλλους τομείς θέλουμε τη συνεργασία και τη συνεχή δέσμευση των κρατών μελών. Αλλά και τη δέσμευση του Κοινοβουλίου και των άλλων οργάνων. Πρέπει να αναφερούμε σε τακτά διαστήματα το έργο μας, ώστε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή χρήση όλων των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας. Διάλογο για, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, διμερείς βοήθεια, δράσεις μας σε πολυμερή βήματα συζήτηση και ούτω καθεξής. Και θα πρέπει βέβαια να επανεξετάζουμε και την πολιτική μας και τη στρατηγική μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήταν χρήσιμο αυτό. Θα ξεκινήσω λοιπόν επισήμω διαβουλεύσεις για την ανάπτυξη μια νέα στρατηγική για τα ανθρώπινα δικαιώματα φέτο. Αξιότιμοι βουλευτέ, αγαπητοί φίλοι, η Έλληνο Ρούσβελτ έλεγε ότι είναι ε, πολύ σημαντικό να ανάψει μάλλον ε, κανείς ένα κλειδί, ένα κερί, αντί να ε, το σκοτάδι. Νομίζω λοιπόν ότι και εμείς ε, μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα όλοι μαζί, βελτιστοποιώντας και μεγιστοποιώντας τις δυνατότητες ε, της νέας στρατικής της Λισαβόνας και βασιζόμαστε στη δική σας υποστήριξη. Gracias. Gracias, señora Τώρα θα δώσουμε το λόγο πρώτα στους ομιλητές που παρεμβαίνουν εξ ονόματος των ε, κοινοβουλευτικών ομάδων. Και πρώτα για 1,5 λεπτό θα μιλήσει ο κύριος Τόκης εξ ονόματος του Έλκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και είμαι σχεδόν εισηγητής εν ονόματι ε, του ΕΛΚ και συντονιστής της πολιτικής μου ομάδος. Οπότε θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την κυρία Χαουτάλα για τη θαυμάσια εργασία που έκανε με την έκθεση αυτή, διότι η ε, ψηφοφορία στην αρμόδια επιτροπή απέδειξε ότι ε, υπάρχει σύγκληση απόψεων μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ομάδων, διότι τα ανθρώπινα δικαιώματα μας ενδιαφέρουν όλους και γι' αυτό καταλήξαμε σε καλές συμβιβαστικές λύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη κατάρτισε μηχανισμούς πολύ σημαντικούς και όπως τόνισα και στις προηγούμενες συζητήσεις πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα επιτύχουμε καλύτερη εφαρμογή των ισχυουσών κατευθυντηρίων γραμμών ότι θα αξιολογήσουμε τις πολιτικές που εφαρμόζονται και ε, ε, θα ρίνω τα κράτη-μέλη να δείξουν πιο ισχυρή πολιτική βούληση για να υπεραμπηθούν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως άλλωστε το τονίζει και η έκθεση διότι ε, εφόσον ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας πρέπει η προστασία των δικαιωμάτων των προσπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να εξασφαλιστεί και προς τρίτες χώρες και σε όλα τα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως κατά τρόπον ώστε να αυξηθεί η συνεκτικότητα ε, σε όλα τα επίπεδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος των Σοσιαλιστών έχει το λόγο για δύο λεπτά η κυρία Βερονίκη Ντοκεζέρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί πολλέ προσδοκίε στι γειτονικέ χώρε, διότι συνεχίζει να σαρκώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πολλέ φορέ όμω διαψεύδονται οι ελπίδε αυτέ, διότι δεν υπάρχουν πολλά τα αποτελέσματα που να συνοδεύουν τα γενναιόδωρα λόγια μα. Βέβαια, με τη βία δεν γίνεται τίποτα. Μόνο με το χρόνο και μέσω συνεκτικών, συνεπών πολιτικών, οι οποίε βασίζονται στην κοινωνία των πολιτών και στι δημοκρατικέ αναδυόμενε δυνάμει. Μόνο έτσι μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο, ιδίω όταν ε, πρόκειται για ε, δικτατορίε ή για διαφθαρμένα ε, καθεστώτα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στη διάθεσή τη ένα καταπληκτικό εργαλείο, δηλαδή την εκλογική παρατήρηση. Αυτό το οποίο όμως εμείς παρατηρούμε στις διάφορες αποστολές εκλογικής παρατήρησης είναι ότι σε πολλές, σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι εκλογές και πολλές φορές είναι ανεπαρκείς και νοθευμένες. Αλλά δεν σημαίνει αυτό κατά ανάγκη ότι από το Συμβούλιο ή από τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ υπάρχει συντονισμένη αντίδραση η οποία γίνεται ακουστή. Και όταν ε, τελικά οι πολιτικοί κάνουν απάτες ε, μετά ε, τις εκλογές ουσιαστικά καταστέλουν και καταπιέζουν τους πολίτες και εμείς νομιμοποιούμε με κάποιες μελέτες ε, κάποια διαφθαρμένα καθεστώτα. Έτσι είναι λίγο μια στρεβλή ε, συνέπεια των εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας. Εγώ υποστηρίζω αυτό το εργαλείο της εκλογικής παρατήρησης, επαναλαμβάνω, αλλά θα ήθελα να υπάρχει, κυρία Άστρο, μια στρατηγική αντίδραση, η οποία θα είναι λίγο πιο ε, προβεβλημένη και πιο ακουστή γενικότερα. Δεν σας άκουσα, μάλλον δεν θέλω να σας αναφέρω τώρα παραδείγματα, αλλά είναι πολλά αυτά τα παραδείγματα. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ντεκάιζερ εκ μέρους των Φιλελευθέρων για ένα λεπτό συνάδελφος Κάζακ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Άστον, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, Προσπαθούμε ε, να ρυθμίσουμε το εμπόριο εργαλείων βασανιστήριων για τιμωρία και οι διεθνείς σχέσεις δεν μπορούν να βασιστούν στην καταπολέμηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχει ένας μακρύς κανόνα, κατάλογος των εργαλείων αυτών και δεν φτάνει να τον ενημερώσουμε. Θα πρέπει συγχρόνως να ε, εξετάσουμε ποια από τα ε, προϊόντα αυτά απαγορεύονται και επίσης πώς εφαρμόζεται ο κανονισμός 1236 διότι ενδέχεται να μην υπάρχουν επαρκές πληροφορίες η πολιτική θέληση δεν υπήρξε στο παρελθόν τώρα όμως δεν έχουμε δικαιολογία και ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, δημοσιεύσει μια λεπτομερή έκθεση για το εμπόριο εργαλείων βασανιστήριων και να βασιστεί στην παραγωγή η οποία είναι αντίθετη προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εξ των Πρασίνων, το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Λόχμπιλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Άστον. Δεν πρέπει να συνεχίσουμε τα βασανιστήρια ε, των κόσμων και πολλά γίνονται. Υπάρχει κατευθυντήρια γραμμή ε, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ενάντια στα βασανιστήρια και ε, θα πρέπει στο μέλλον να τονίσουμε ότι τα απαγορευτικά μέτρα παραγωγής εργαλείων βασανιστήριων έχουν κενά και αυτό αποβλέπει και το ψήφισμα το οποίο θα υπερψηφιστεί αύριο. Δεν πρέπει όμως να ε, ε, καταλήψουμε την προσπάθεια να ονοματίσουμε τα κράτη τα οποία ε, συμμετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες διότι η έκθεση της Lady Ashton αποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζεται εκ των έξω και βλέπουμε πως η ίδια παρακάμπτει τα, τις προδιαγραφές προστασίας. Πρέπει λοιπόν και εμείς να κατακρίνουμε τις δικές μας πράξεις και να μην ευθυνόμαστε μόνο και να στρεφόμαστε στις εξωτερικές πολιτικές για να μπορούσαμε να είμαστε αξιόπιστοι. Επίσης τώρα, η κυρία ε, ε, δείχνει την ε, μπλε κάρτα, τη γαλάζια κάρτα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτή η κάρτα. Σημαίνει ότι θέλετε να υποβάλλετε μία ερώτηση προς την κυρία Λόχμπίλερ, έτσι να το ερμηνεύσω. Ή θέλετε να εγγραφείτε για τις παρεμβάσεις ενός λεπτού. Α, αυτό ισχύει, εντάξει. Εξ των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών για δύο λεπτά έχει το λόγο ο δόκτωρ Τάνοκ. Η ιστορία μας διδάσκει ότι πρέπει να τηρούνται τα υψηλά πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε περήφανοι για το τι έχει πετύχει σε αυτό το τομέα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά γι' αυτό το λόγο πρέπει να ενισχύσουν τις προσπάθειές μας να προβάλλουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις περιοχές του κόσμου όπου καταπατώνται και αγνοούνται. Παραδείγματος χάρη ομοφυλόφιλοι, οι μυχοί, οι μιχαλίδες και άλλοι άνθρωποι ε, θανατώνονται σε τακτική βάση ή αυτά που συμβαίνουν στην Κορέα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης για εκείνους που προσπαθούν να ξεφύγουν από αυτόν τον εφιάλτη. Ας πάρουμε τη Βυρμανία όπου η στρατιωτική στρατοπεδα συγκεντρωσης για εκεινου που τρομοκρατεί τον πληθυσμό και τη Βενεζουέλα της οποίας ο ηγέτης Λούγκο Τσάβες έχει κλείσει και φημώσει τα μέσα ενημέρωσης Δώσαμε πέρσι το βραβείο Ζαχάροφ στον οργανισμό, στην οργάνωση που αγωνίζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία και που αγωνίζεται κυρίως κατά τις δολοφονίες δημοσιογράφων. Δεν πρέπει βεβαίως το μόνο γνώμο, ο μόνος γνώμονας για τη σχέση με τις διάφορες χώρες δεν πρέπει να είναι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Κίνα όμως ε, που είναι πολύ καλός ε, εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθεί να παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το ίδιο ισχύει και στο Πακιστάν. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ρεαλιστές για αυτό που μπορούμε να πετύχουμε. Να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας να πείσουμε τους άλλους για τη σημασία των δημοκρατικών μας αξιών που τόσο πολλοί μας έχουν υπηρετήσει το να απαγορεύσουμε το εμπόριο σε εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για βασανιστήρια είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δείξει ότι αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Τανόκ εξ ονόματος της ε, Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς για 1,5 λεπτό. Έχει το λόγο κυρία Βαριζά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναγνωρίζονται πάνω απ' όλα από τις πράξεις τους. Είναι όλοι εκείνοι και εκείνες που με εκείνη τη ζωή τους αγωνίζονται σε ολόκληρο τον κόσμο για να εφαρμόσουν και να προασπίσουν όλα τα δικαιώματα έτσι όπως προκύπτουν από την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τα κείμενα που την συμπλήρωσαν. Ε, εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτή την πρόταση της έκθεσης η αντίληψή μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να είναι εκείνη των Ηνωμένων Εθνών. Πρέπει να προασπίζουμε μία μοναδική αντιμετώπιση και προσέγγιση στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οικουμενική σε ολόκληρο τον κόσμο, αδιέρετη, δηλαδή όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να προστατεύονται με, με ισότιμο τρόπο, χωρίς να αντικρούν τα μέντα εδέ, είτε πρόκειται για πολιτικά, αστικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και άλλα δικαιώματα και πολιτιστικά δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει μια σειρά από μέσα σε αυτού του τομεί και είμαι ευτυχή ε, που τα αναφέρει όλα η έκθεση λαμβάνοντας υπόψη και τις νέες αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστώ λοιπόν την κυρία Ούταλα για την ποιότητα της έκθεσής της και τον τρόπο με τον οποίο δέχθηκε να συνεργαστεί μαζί μας. Η έκθεση αυτά είναι αρκετά επικριτική σε ό,τι αφορά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι γνωρίζουμε ότι μεταξύ των λόγων και των πράξεων υπάρχει μεγάλη απόσταση. Τα οικονομικά και διπλωματικά συμφέροντα έχουν το προβάδισμα σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και υποφέρουν άνθρωποι γι' αυτό. Η πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών εφαρμόζει μεταβλητή γεωμετρία. Για μένα αυτό είναι κάτι το απαράδεκτο με αυτή την έκθεση που πέρα του γεγονό του καταδικάζει κάθε βία κατά των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, διαγράφουμε διάφορε κατευθύνσει που θα πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε να μπορέσει να ενισχύσει την αξιοπιστία τη Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε μέσα. Ναι κυρία Άστον, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε σε αυτόν τον τομέα. Η προηγούμενη συζήτηση μας το έδειξε. Όπως και εκείνη που θα λάβει χώρα αύριο το απόγευμα για τη Λιβύη. Θα μας το δείξει επίσης. Όπως και η πολιτική που θα ε, ε, υιοθετηθεί για τις πωλήσει εργαλείων για ε, βασανιστήρια που, στις οποίες προβαίνουν ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Εξ της Ελευθερίας και Δημοκρατίας για 1,5 λεπτό έχει το λόγο ο κύριος Κάμπελ Μπάνκμ. Κύριε Πρόεδρε Βαρόνι, όλοι είμαστε υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βεβαίως όλα αυτά έχουν εγγραφεί στη Μάγνα Κάρτα του 1215 και άλλων μεταγενέστερων νομοθετικών εγγράφων καθώς και εγγράφων και συμφωνιών που ανέκυψαν μετά από τον πόλεμο. Δυστυχώς όμως υπάρχουν καιροσκόποι που ε, δυστυχώς ε, αντιπροβάλλουν κάτι το εντελώς διαφορετικό. Και από ό,τι φαίνεται θα πρέπει να δούμε κατά πόσο πρέπει να επιτρέψουμε ακόμα και στους φυλακισμένους να ψηφίζουν. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε τους ε, πολίτες, όχι τους ε, τρομοκράτες, τους εγκληματίες και αυτούς που παραβαίνουν το νόμο. Μπορεί οποιοδήποτε δικαστήριο να ζητήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο να ζητήσουμε τον, την ψήφο από φυλακισμένους και καταδικασμένους, όπως ισχύει με έναν εγκληματία στη δική μου εκλογική περιφέρεια μπορούμε να ζητήσουμε την ψήφο της Rosie West που ήταν ε, κατά δολοφόνος ή άλλων δολοφόνων στην Ευρώπη. Ποιους θα υποστηρίξουν ακόμα και αν ψηφίσουν. Αυτοί όμως οι φυλακισμένοι θα μπορούσαν να ψηφίσουν σε τοπικό επίπεδο και να ε, κατάγουν συντριπτική νίκη. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε λοιπόν την ψήφο των εγκληματιών και των πρώην ε, φυλακιστέντων. Δεν μπορούν να συμμετέχουν στην πολιτική διαδικασία και στην ε, πολιτική δημοκρατία τη στιγμή που προκάλεσαν θύματα. Πού έγκυται η ανθρώπινη ευθύνη. Νομίζω ότι όπως και το ευρώ έτσι και το κοινό νόμισμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει υποβαθμιστεί. Πρέπει να επανέλθουμε στην κοινή λογική. Από τους μη εγγεγραμμένους, η κυρία Σίνκλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως τονίζει η συγγήτρια, με βάση τη διακρίση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλοι έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν ως οικουμενικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση φαίνεται να σκέφτεται διαφορετικά επειδή προβάλλει ορισμένα ανθρώπινα δικαιώματα σε βάρος άλλων. Τα δικαιώματα των ταξιδιωτών παραδείγματο χάρη και στη δική μου εκλογική περιφέρεια πιστεύουν οι κάτοικοι ότι δεν γίνονται σεβαστά όλα τους τα δικαιώματα. Πρέπει λοιπόν να καταβάλουμε προσπάθειες για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα των επομένων γενιών. Στη δική μου τοπική κοινότητα γίνονται προσπάθειες ώστε όλοι να τηρούν τις υποχρεώσεις τους και να προστατεύουν τα δικαιώματα πολιτών, πολιτών οι οποίοι το μόνο που θέλουν είναι να προστατεύσουν τα δικαιώματα τα δικά τους και της οικογένειας τους. Συμφωνώ με την εισηγήτρια. Πρέπει οπωσδήποτε να προστατεύσουμε και να στηρίξουμε εκείνους που αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Γάνα, στη, Γά, ε, στη Γάζα, στην Κύπρο και παντού. Αλλά αυτό που προσπαθώ να πω είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα κινδυνεύουν, κινδυνεύουν παντού είναι όμως πολύτιμα και πρέπει να προστατεύονται και στη δική μας χώρα και παντού σε ολόκληρο τον κόσμο. Μου κοινοποιούν οι διερμηνείς ότι μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα και είναι αδύνατο να περάσουν τα μηνύματά σας με αυτό το ρυθμό που μιλάτε. Να το έχετε υπόψη σοβαρά αυτό, γιατί διαφορετικά οι διερμηνείς δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Μας το κοινοποιούν και να το λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη. Δεν μπορεί μέσα σε ένα λεπτό να θέλετε να διαβάσετε πέντε σελίδες ο καθένας. Πρέπει να είσαστε λογικοί. Τελειώσαμε λοιπόν με τον γύρο αυτών των ομιλητών και περνάμε στους ομιλητές που δεν μιλούν εξ ονόματος της πολιτικής τους ομάδας. Ο κύριος Γκρέις έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξότιμοι βουλευτέ, ε, πρέπει βέβαια να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι σημαντικό τμήμα τη εθνική πολιτική, ιδίω τώρα που έχουμε νέε αρμοδιότητε βάσει τη τήξη Λισαβόνα. Η έκθεση που μα ε, παρουσιάστηκε είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εγγραφό. Δεν μπορούμε ε, τώρα να αναφερθούμε σε όλα τα στοιχεία, όλα τα στοιχεία της έκθεσης αυτής. Θα ήθελα να εκφράσω καταρχήν την ε, ικανοποίησή μου που έχουμε αυτόν το διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν είναι πάρα πολύ επιτυχής, ιδίως όσον αφορά τις γειτονικέ χώρες και τις ε, χώρες της ε, Ανατολικής γιατί σχέση Στρέφουμε προς εμάς, λέει διάστον, και προς τον Επίτροπο Φίλερ, θα πρέπει να δώσουμε κατά τον περισσότερα ενάβσματα για να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπως είπε η θα πρέπει να αποστείλουμε ευφυή μηνύματα και να κατατρέξουμε ή οικονομικά ή πολιτικά οποιοδήποτε καταπάτησε των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά τα στοιχεία συμπεριλαμβάνονται και στην έξι κυρία Σαουτάλα. Και θα ήθελα να τονίσω ότι το βραβείο Σαχάροφ που δίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα οδηγήσει στην υποστήριξη αυτών που βραβεύονται από όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν ίσως να χρησιμοποιήσουμε αυτό το δίκτυο δικηγόρων. Είχαμε κάποιες ε, διαδηλώσεις στον, ε, στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη για την έλλειψη ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ρωσία και δεν αντιδράσαμε εμείς. Και ένας από τους που είχε στραφεί για μας για να τους υποστηρίξουμε ήταν ε, ένας βραβευμένος με το βραβείο Ζαχάροφ. Θα πρέπει τώρα να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας καλύτερα για να προσπίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Απευθύνομαι σε όλους τους συναδέλφους. Θα ήθελα να σας κάνω μία στεναρή έκκληση να αρκείστε στο χρόνο ομιλία σας. Γιατί δεν θέλω να σας διακόψω ή να σας διακόπτω, αλλά αναγκάζομαι να το κάνω. Γιατί είδατε ότι χτες κατά τη νυχτερινή ολομέλεια υπερβήκαμε τις 12 κατά πολύ. Θα πρέπει λοιπόν να αρχίσω να σας διακόπτω. Το λόγο έχει τώρα για δύο λεπτά ο συνάδελφος Βιτόριο Πρόντι. Ευχαριστώ Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και την Αντιπρόεδρο, την Βαρόνι Άστον. Οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαδραματίζουν ε, ζωτικό ρόλο και θέτουν σε κίνδυνο και τη δική τους ζωή. Η τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι μία από τις θεμέλιες λήθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οδήγησε στην οικοδόμησή της. Γι' αυτό θα πρέπει να επιμένουμε στην τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχοντας μία ολιστική θεώρηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια Χαουτάλα για την εξαιρετική της εργασία. Και οι σοσιαλιστές και δημοκράτες συνεισέφεραν σε αυτή την εργασία. Θα πρέπει όμως να κινηθούμε πέραν της έκθεσης, θα πρέπει να αναλάβουμε σαφώς την ευθύνη μας και να ασχοληθούμε πιο σοβαρά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, διότι πρόκειται για ένα περίπλοκο φαινόμενο που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε σφαιρικά. Είμαι πεπισμένος ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και την, το δικαίωμα στους πρόσβασης στους φυσικούς πόρους, το δικαίωμα σε συστήματα υγείας, στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στην πληροφόρηση. Με τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, θεωρώ ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έτσι ώστε να προβάλλουμε το έργο μας σε αυτό το τομέα. Η κυρία Άστον τόνισε αυτή την πτυχή του θέματος ως προς τις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε καθημερινά προκλήσεις, τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στεναρά, διότι είμαστε πρωταγωνιστές στο διεθνές προσκήνιο. Η κυρία Όγιουλαντ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Θα ήθελα να υπογραμμίσω με τη σειρά μου τις, τις ευχαριστίες μου προς τη Λέδη Άστον και τις πολύ σαφείς και ξεκάθαρες θέσεις που μας παρουσίασε. Στην έκθεση της συναδέλφου Χάουταλα έχει τονιστεί κάποιο συγκεκριμένο σημείο. Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η υπόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διεθνείς συμφωνίες επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει σαν προϋπόθεση την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αν δεν θέλει να είναι κενέ λέξεις τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει με συνέπεια να εφαρμόζει την πολιτική τη η Ευρωπαϊκή Ένωση και να καλεί τα κράτη-μέλη να αναλάβουν πιο συντονισμένη δράση έναντι τρίτων χωρών. Έχουμε οικονομικού και άλλου μοχλου που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν μέσα πίεση για την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Διότι αλλιώ με αυτόν τον τρόπο οι χώρε που παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα θα δουν τα συμφέροντά τους να πλήττονται. Εάν δεν γίνει αυτό, οι χώρες αυτές θα συνεχίζουν να συμπεριφέρονται έτσι όπως συμπεριφέρονται τώρα. Τα οικονομικά μας συμφέροντα δεν πρέπει να θεωρηθούν πιο σημαντικά από τις αξίες που εκφράζει στο σύνολό της Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό λοιπόν την Λέδη Άστο να μας αναφέρει τι μέτρα σκοπεύει να λάβει. Ευχαριστώ, που σας, ευχαριστώ που σας διάκοψα. Ο κύριος Αρνέσκη είναι ο επόμενος ομιλητής. pani przewodnicząca! inteligencja. θα ήθελα να πω προς την ύπατη εκπρόσωπο ότι είμαστε ευφυή όντα και αυτό δείχνει ότι πολλές φορές δεν τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι αξίες μας και εμείς το παραγνωρίζουμε. Αυτό που έχει σημασία και μας ανησυχεί είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο και η Επιτροπή βλέπουν υπό διαφορετική οπτική γωνία το ίδιο θέμα όταν παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα σε χώρες που δεν παρουσιάζουν μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρον ή οικονομικό ενδιαφέρον για τα περισσότερα κράτη-μέλη. Σε αυτή την περίπτωση, οι οικονομικές αναλύσεις είναι εντελώς διαφορετικές και εντελώς διαφορετική η θεώρηση αυτών των παραβιάσεων. Όταν παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα σε χώρες με τις οποίες έχουμε μεγάλες εμπορικές συναλλαγές, έφνης φαίνεται ότι σιωπούν οι πάντες. Αυτή, θα πρέπει, αυτή η τακτική θα πρέπει να σταματήσει. Η κυρία Αντρικιένε έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω ότι η έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο είναι ιδιαίτερα σημαντική και καλύπτει πάρα πολύ τα περισσότερα από τα σημαντικά θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει ότι η έκθεση περιγράφει τις ενέργειες Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά επανάληψη έχει διατυπώσει συστάσει λέγοντα ότι πρέπει να αναπτύξει δείκτε και στοχοδείκτε ειδικότερα το, το Συμβούλιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένωσης ώστε να μπορεί να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σχετικά θέλω να αναφερθώ και στην πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα στοιχεία και τις πληροφορίες που διαθέτουν το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτι που παρέμεινε περιορισμένο μέχρι στιγμή, παρόλε πολλαπλέ πολλαπλές για αυτό το θέμα του Κοινοβουλίου η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί. Θα αναφέρω το διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα σαν παράδειγμα που διενεργούνται με τι αρχέ διαφόρων χωρών. Το Συμβούλιο είχε μια σειρά από ε, συζητήσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη Ρωσία. Γνωρίζουμε πολύ καλά ποια είναι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία. Οι ε, δημοσιογράφων, ο τρόπος αντιμετώπισης των δίθεν ε, τρομοκρατών σε ορισμένες περιοχές κλπ. Θα θέλουμε όμως να ξέρουμε ποια ήταν η αντίδραση των Ρώσων που ήταν παρόντε στο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρόκειται να, ληφθούν, να γίνουν κάποιες ενέργειες σχετικά πέρασε ο χρόνος μου, το ξέρω. Αλλά θα ήθελα απλώ να πω ότι κατανοώ απόλυτα ότι εντάσσονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θέματα της ασφάλειας μπορούν να θεωρηθούν ενδεχομένω σαν κάτι σαν τομέα, που υπάρχει στον τομέα της ασφάλειας, αλλά κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Χαουτάλα για το πώς αντιμετώπισε το θέμα στην Υποεπιτροπή, καθώς και την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, σε σχέση με τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις υποχρεώσεις. Προωθούμε τον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες, αλλά ο διάλογος δεν είναι αυτός σκοπός. Γι' αυτό θα ήθελα να αναγνωρίσω τις συζητήσεις της ΥΠΑ της εκπροσώπου, έτσι ώστε να διοχετεύσουμε αυτές τις δράσεις στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Συζητάμε νέες ιδέες, έτσι ώστε να έχουμε μία ε, οριζόντια αντιμετώπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να έχουμε μια υπηρεσία ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις αντιπροσωπίες μας. Ίσως αυτά να εντάσσονται σε ένα κείμενο νομοθετικού περιεχομένου, ίσως όχι. Παρακαλώ να επιβραδύνετε, λέει ο Πρόεδρος. Δεν θα ήθελα να υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις στη σύσταση αυτών των υπηρεσιών παντού, θα πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη ότι αυτά είναι εύκολα, υπάρχουν εύκολα επί χάρτου, αλλά δεν σημαίνει ότι τίθενται σε εφαρμογή. Νομίζω ότι με αυτή τη νέα υπηρεσία θέλει το Κοινοβούλιο να συνεργαστεί μαζί της έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε την άκρη και αυτού του μύτου. Ευχαριστούμε κύριε Χάουιτ. Το λόγο έχει η κυρία Σάκε για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Άστον και θέλω να πω ότι ήταν πάρα πολύ ωραία η συνεργασία με τους συναδέλφους που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω ότι έφτασε η στιγμή να δούμε ποιες είναι οι υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο. Εμεί έχουμε συντάξει μια γραπτή διακήρυξη υπέρ των Ιρανών και του αγώνα τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συναντηθήκαμε με τον Ζενιά Σαντάν που είναι ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θέλει να εμποδίσει την, θα, την θανατική καταδίκη για τα παιδιά. Μια πρακτική που πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει. Χρειάζεται περισσότερο συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δικαιούνται ευρύτερη και ολοκληρωμένη προσέγγιση. Υπάρχουν δυστυχώ γεωγραφικέ περιοχέ στι οποίε εξακολουθούν να παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπω τα δικαιώματα των γυναικών, το δικαίωμα τη ελευθερία τη έκφραση που διαρκώ παραβιάζονται. Το καθεστώ του Ιράν είναι ένα παράδειγμα όλων αυτών των παραβιάσεων. Η, δυστυχώς η, Ευρω... παγκόσμια κοινότητα στην περίπτωση του Ιράν δεν ασχολείται με τίποτε άλλο παρά μόνο με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις από τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά φοβάμαι ότι δεν θα έχουν και τόσο σημαντικά πρακτικά αποτελέσματα. Πρέπει ο λαός πρέπει οι κάτοικοι του Ιράν να έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως και οι λαοί σε άλλες περιοχές του κόσμου. Έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που έγιναν προεδρικές εκλογές στο Ιράν με αποτέλεσμα να ασκείται ακόμα περισσότερη βία και καταπίεση εναντίον του λαού. Η αντιπολίτευση πλέον έχει φημωθεί πλήρως πολλοί προσπάθησαν να φύγουν και να έρθουν στην Ευρώπη και πιστεύω ότι πρέπει να τους υποδεχθούμε διότι θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να καθορίσουμε την ορθή πολιτική που θα πρέπει να ακολουθήσουμε σε σχέση με αυτή τη χώρα. Ο κύριος Μιγκάλσκι έχει το λόγο για ένα λεπτό. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Είμαι πολύ ευτυχής που η Λέδη Άστον έμεινε μαζί μας και παρακολουθεί αυτή τη συζήτηση. Το θεωρώ αυτό ότι σαν έκφραση ενδιαφέροντός της για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μπορεί να διαφέρουμε από σε κοινωνικά και γεωπολιτικά θέματα στην Ευρώπη, σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, μιλάμε με μία φωνή, παρόλες κάποιες διαφ... παρόλο το γεγονός ότι προερχόμαστε από διαφορετικές χώρες και από διαφορετικά κόμματα. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας ενώνει. Είναι παράδοξο λοιπόν πιστεύω ότι δεν έχουμε ακόμα καταφέρει να, ε, να υπερασπιστούμε εκείνους τους οποίους απονέμουμε βραβεία. Το βραβείο Οι ε, αποδέκτες του βραβείου Ζαχάροφ έχουν δεχθεί ε, επιθέσεις διώκονται την ίδια τους τη χώρα. Οι βραβευθέντες με το περσινό βραβείο και εκείνοι αντιμετωπίζουν την, την ίδια συμπεριφορά από τις αρχές της χώρας τους. Πρέπει λοιπόν να προσφέρουμε προστασία σε όλους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα σε εκείνους στους οποίους έχουμε βραβ... απονείμει τα βραβεία μας, το βραβείο μας. Ε, Ο κύριος Κασμάρεκ έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω προς την ύπατη εκπρόσωπο ότι μιλάμε για την τήρηση και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρόκειται για μια καθολική αξία και δεν μπορούμε παρά να την προωθήσουμε ανά τον κόσμο. Όμως, η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε χώρες που απειλούνται, όπου υπάρχει ιδιαίτερη απειλή, εκεί θα πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο το θέμα των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γίνονται θύματα μιας ε, πάγιας και μόνιμης απειλής από το κράτος. Γίνονται ε, παράνομες κρατήσεις, φυλακίσεις, βασανιστήρια. Γι' αυτό θα πρέπει να βοηθήσουμε όλους εκείνους που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι μέρος των μόνιμων υποχρεώσεών μας. Πρόκειται για μια, κίνηση συμβολικής και ηθικής αξίας θα πρέπει όμως να υπάρξει και μία υλοποίηση προγράμματος από πολιτικής και διπλωματικής πλευράς, διότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πεθαίνουν πολλές φορές μέσα σε φυλακές ή δολοφονούνται. Αύριο θα αναφερθούμε στο θάνατο ε, ενός από τους υπερασπιστές και είναι κάτι που δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Το λόγο έχει η κυρία Μαρία Μουνή για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στα, στο εμπόριο εργαλείων βασανιστήριων που θα ψηφίσουμε. Θα πρέπει να δούμε ορισμένα απτά παραδείγματα έτσι ώστε να εφαρμόσουμε καλύτερα τα διεθνή ψηφίσματα. Θα ήθελα να συγχαρώ τα επτά κράτη τα οποία συντάσσουν ετήσιες εκθέσεις για το εμπόριο αυτών των εργαλείων βασανιστήριων. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους και να, είμαστε, να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς αυτό το θέμα. Το εμπόριο αυτό απαγορεύεται, όπως αναφέρεται στο παράρτημα 2, καθώς και ε, εργαλεία που οδηγούν σε βασανιστήρια, τα οποία θα πρέπει να προσαρτηθούν στη, στον κατάλογο. Αυτό θα προτείνω στην Ισπανική Προεδρία, έτσι ώστε να μην είναι δυνατόν να γίνεται εμπόριο αυτών των εργαλείων. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποστείλει ένα μήνυμα ότι δεν μπορούν να προωθηθούν ή να εμπορεύονται αυτά τα εργαλεία τη στιγμή που διασαλεύεται η δημόσια τάξη, η ασφάλεια, όπως πολλές ε, φορές προβάλλεται από κατασταλτικές χώρες. Ευχαριστούμε. Βοησχεχόφσκι για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω κάποιες σκέψεις όσον αφορά τον πλανοσμό για την απαγόρευση του εμπορίου εργαλείων βασαστηρίων. Αυτά τα εργαλεία τα βλέπουμε συχνά σε μουσεία, αλλά δεν είναι πράγματα που ανήκουν μόνο στην, στα μουσεία. Είναι εργαλεία που χρησιμοποιούνται και σήμερα. Τα βασανιστήρια γίνονται ε, όχι μόνο ανά τον κόσμο, αλλά και σε ορισμένε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας είναι να καταπολεμήσουμε τα βασανιστήρια η οποιαδήποτε μορφή και η απαγόρευση αυτή των, ε, ε, του εμπορίου των εργαλείων βασανιστήριων θα πρέπει να εφαρμοστεί όσο δυνατόν ευρύτερα. Δεν μπορούμε να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Οι άνθρωποι που εκτίθεται σε βασανιστήρια παραδέχονται οτιδήποτε βέβαια, ομολογούν τα πάντα και οι πραγματικοί δράστες ε, δεν ε, τιμωρούνται, δεν συλλαμβάνονται καν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ένα μισό λεπτό. Η κυρία Κίνγκα Γκάλ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, θα πρέπει πραγματικά να αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία στους πρόσφυστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να αναγνωρίσουμε το έργο τους και αυτό όχι μόνο εκ των υστέρων, είναι κατά γνώμη πάρα πολύ σημαντικό το Κοινοβούλιο να εκφράσει την άποψή του εδώ και συγχαίρω την εισηγήτρια για την έκθεση πρωτοβουλία που υπέβαλε. Πρόκειται για μια πάρα πολύ καλή εργασία η οποία απαριθμεί ακριβώ τι χρειάζεται. Και γι' αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε πιο προσπάθεια, ούτω ώστε αποτελεσματικά και γλίγορα να χορηγείται βοήθεια στους ανθρώπους αυτούς. Είναι και τα δύο σημαντικά. Και η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, οι προσπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διακυβεύουν την ίδια τη ζωή τους. είναι σημαντικό να έχουμε ένα καλά, μια καλά δομημένη υπηρεσία εξωτερικής δράσης που να ε, μπορούν να εξαρθούν και τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως είπαν και διάφορα άλλοι συνάδελφοι. Εσείς στην Κομισιόν είσαστε τώρα εκείνη που έχετε τον μπαλάκι στα χέρια σας για να αναλάβετε ε, συγκεκριμένα πρακτικά βήματα. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό ο κύριος Ζένκε. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. όταν ε, συζητάμε τα ανθρώπινα δικαιώματα χρησιμοποιούμε πολλούς ε, μεγαλόπνοες ιδέες και λέξεις που παρουσιάζουμε χωρίς να έχουμε τις ανάλογες πράξεις που να ακολουθήσουν. Γιατί αυτές οι εκθέσεις και οι ομιλίες ε, της, ε, του Κοινοβουλίου που λένε ότι θα πρέπει να λάβει πιο συγκεκριμένα μέτρα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικά. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τους πρόσπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πολύ καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Έχουμε αυτούς τους θαυμάσια ε, θαραλέους ανθρώπους που θα πρέπει πραγματικά να μην τους αφήνουμε στη μοίρα τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα προετοιμάζει ένα κώδικα θεωρήσεων διαβατηρίων για την κοινότητα και θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω κατά πόσον αυτός ο κώδικας για τις θεωρίες διαβατηρίων θα διακανονίσει το θέμα της χορήγησης ε, θεωρήσεων στους προασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν απειλείται η ζωή τους. Εκτός αυτού, ε, θα υπάρχουν υπεύθυνοι για τις θεωρήσεις στα γραφεία της εξωτερικής δράσης. Ευχαριστώ προς διακόπτη. Ο κ. Πρωτακίεβιτς έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Και λέει Άστον, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να αρχίσω ευχαριστώντας την εισηγήτρια για το έργο που επετέλεσε. Με ικανοποίηση άκουσα αυτά που είπε η Λέδη Άστον ότι θα πρέπει η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να είναι κύρια μας προτεραιότητα. Απ' την άλλη μεριά με ανησυχεί η πολύ αδρανής και παθητική μας στάση όσον αφορά την ε, καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παραδείγματος χάρη στη Ρωσία ή στη Λευκορωσία, όπου εξακολουθεί να επιβάλλεται η θανατική ποινή, επιβαλλεται η θενατικη άνθρωποι φυλακίζονται επί χρόνια και ότι αν είναι κανένα μέλος μιας μη κυβερνητικής ε, κυβέρνησης σημαίνει ότι διώκεται. Πολλά ακόμα θα πρέπει να γίνουν για να βελτιώσουμε την πολιτική αυτή και θα πρέπει να είναι γρήγορη και αποτελεσματική η οποιαδήποτε δράση, κυρία Επίτροπε, ιδίω όταν τα θεσμικά όργανα δεν μπορούν να κάνουν πολλά, είναι πολύ αδρανή η Ισπανική Προεδρία νομίζω ότι πραγματικά αδράνησε από αυτού. Ελπίζω στην αυριανή συζήτηση να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε την προσοχή μα περισσότερο στην κατάσταση στη Ρωσία. Γιατί δεν χρειάζεται να λέμε μόνο κάτι για αυτό που γίνεται στη Λευκορωσία, πρέπει να πράξουμε κιόλα. Τελειώσαμε τον κύριο Πρασίεβιτς, τον κατάλογο των ομιλητών και θα περάσουμε στον γύρο του Catch the Eye. Είχαμε ένα πρόβλημα εδώ. Δηλαδή συνήθως πέντε συνάδελφοι πρέπει να ζητήσουν το λόγο. Έχω δεκαπέντε όμως καταγράψει. Και συνήθως είμαι πιο ευέλικτος. Σήμερα όμως δυστυχώς δεν μπορώ να είμαι ευέλικτος και δεν θα δώσω σε κανέναν το λόγο που ε, έλειπε κατά διάρκεια της συζήτησης και τώρα ήρθαν τρέχοντας για το Καστιά για να πει κάτι. Αυτό δεν είναι λογικό μου φαίνεται σε αυτές τις περιποθέσεις να σας δώσουμε το λόγο. Λοιπόν, πέντε άτομα θα πάρουν το λόγο με τη σειρά που έχουμε καταγραφεί. Βανέσα πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ολοκληρωμένη και πολύ ενδιαφέρουσα έκθεσή της. Συμφωνώ ότι η στάση Ευρωπαϊκής Ένωσης ως υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνδέεται άμεσα με την εσωτερική αρχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Γι' αυτό υποστηρίζω την έκθεση όταν λέει ότι είναι απαραίτητο να καθιερωθεί μια θέση αξιωματικού <clears throat> συνδέσμου στις αποστολές μας στο εξωτερικό. Η αξιολόγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι απαραίτητη για τις χώρες οι οποίες διατηρούν στενούς εμπορικούς δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανάγκη επιβολής ποινών κυρώσεων σε τρίτες χώρες που παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα είναι και αυτό κάτι που πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε η κυρία Βασίκο Βαβαλόβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέει διάστον σχετικά με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι αναπόσπαστο τμήμα της δημοκρατίας η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο έχει αναλάβει πολλές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις απέναντι στον κόσμο οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διώκονται υφίστανται βία βασανιστήρια κλπ μετά από την ε, θέση της συνθήκη της Λισαβόνας πρέπει να παίζουμε ηγετικό ρόλο μέσω των αντιπροσωπιών μας σε τρίτες χώρες δεν τα έχουμε καταφέρει και τόσο καλά μέχρι στιγμή. Με τι νέε εξουσίε που διαθέτουμε λοιπόν τώρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που διαθέτουμε να βελτιωθεί η κατάσταση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και να προστατεύουν του υπερασπιστέ τη σε όποια χώρα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεία. Θέλουμε εκπροσώπου υψηλού επίπεδου οι οποίοι θα έχουν ω προτεραιότητα την δημοκρατία και τα ε, ε, ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκέρενς έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αν θέλουμε να ακούγει τη φωνή μα σε θέματα προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, α είμαστε άμεμπτοι στη... στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσχώρησε η Ευρωπαϊκή Ένωση ω Ένωση στην ΕΣΔΑ, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κάτι που δείχνει, ελπίζω, την βούληση των 27 να εφαρμόσουν, εφαρμόσουν και όλε τι υποχρεώσει που συνεπάγεται αυτή η Σύμβαση του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να δεσμευθούν η κάθε μία από τι 27 χώρες μέλη να τηρούν και να σέβονται όλες τις αποφάσεις του, του, του Δικαστηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Στρασβούργου. Αναλαμβάνεται λοιπόν να επιβάλλεται σε όλα τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν όλες τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και να με ενημερώσετε σχετικά. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε καταργήσει μία συμπεριφορά που μας δείχνει, που μας κάνει να είμαστε αμήλικτοι, αμήλικτοι απέναντι σε, στις άλλες χώρες, ενώ εμείς ε, μέσα στον δικό μας τον οίκο δεν τηρούμε αυτούς τους κανόνες. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Χαουτάλα για την εξαιρετική έκθεση όπου τονίζει τα μέσα που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδιαίτερα τη ρήτρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προσαρτάται σε κάθε εμπορική συμφωνία. Θα ήθελα να αναφερθώ στις 28 Ιουνίου. Σε μερικές μέρες θα, ε, θα εορταστεί το πραξικόπημα στις, ε, στην Ονδούρα, διότι η βία συνεχίζεται μετά την εγκατάσταση στην εξουσία του Φιρέο Βία κατά των ε, δημοσιογράφων, των ανθρώπων, των γυναικών, πολλοί σκοτώθηκαν και η ΕΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις εμπορικές συμφωνίες σαν να μην είχε γίνει τίποτα. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που διαθέτουμε. Διακόπτεται ο μιλήτρια. Ο κύριος Μπάτεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα Βαρόνι Άστον. Υπάρχει κατάχρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι για το οποίο ελπίζω κάτι θα μπορέσουμε να κάνουμε. Θέλω να την προσοχή σας στις προϋποθέσεις, στις συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική φυλακή του Κορυδαλού. Η μόνη φυλακή όπου εθνικοί, ε, ε, ξένοι αλλοδαποί κρατούνται. Βρετανοί που πολύ συχνά έχουν βρεθεί στον Κορυδαλό. Ένδεκα μήνες ένα, πέρασε ένα συμπολίτη μου στον Κορυδαλό πριν δικαστεί. Τώρα έχει βγει με εγγύηση, αλλά οι συνθήκες, οι συνθήκες ε, ήταν όπως μας είπε αφόρητες. Ο Κορυδαλός έχει κατα... Η φυλακή του Κορυδαλού έχει καταδικαστεί από οργανισμούς όπως την Διεθνή Αμνηστία και άλλες ως η φυλακή με τις χειρότερες συνθήκες στον κόσμο. Παραβιάζει το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Συμφωνείτε μαζί μου. Τελειώσαμε με τις παρεμβάσεις αυτές των συναδέλφων μέσα στα πλαίσια της παρέμβασης του ενός λεπτού. Και έπρεπε να σας διακόψω διότι δεν γινόταν διαφορετικά. Το λόγο έχει η κυρία Άστον για να απαντήσει στις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν από τους βουλευτές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τα μέλη που δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν την παρέμβασή τους βεβαίως τους παρακαλώ να έρθουν σε επαφή μαζί μου για να θέσουν οποιοδήποτε θέμα. Θα ήθελα να πω, καθώς ολοκληρώνεται αυτή η συζήτηση, ότι είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για αυτή την ευκαιρία που είχαμε για μια τέτοια συζήτηση. Πολλές φορές τα σημαντικά θέματα ξεπερνώνται από επίγοντα ζητήματα και είναι σημαντικό ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να εξασφαλίσει ότι παραμένουμε πιστοί στι θεμελιώδει αρχέ που περιέχονται στο Συμβούλιο, στην Συνήθεια τη Αβώνα. Ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα, κράτο δικαίου και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων εκείνων που ανήκουν σε μειονότητες αυτή, αυτός είναι ο γνώμονας, ο που στη, με βάση του οποίου αναπτύσσουμε την εξωτερική μας πολιτική σε όλους τους τομείς. Πολλά, πολλοί συμμετέχοντας μίλησαν για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ανάγκη να συνεχιστεί μαζί τους ο διάλογος. Κατέστησα ήδη σαφές ότι καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να συναντούμε τους ε, ακτιβιστές που αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλα τα μέρη του κόσμου και τους υποδέχομαι με ιδιαίτερη χαρά στο γραφείο μου στις Βρυξέλλες όπως έγινε με κάποιους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αφγανιστάν. Έτσι πρέπει να λειτουργεί η διπλωματική υπηρεσία. Ξέρω ότι ο κ. Δεκάζεκ δεν είναι εδώ αλλά σημείωσε αυτά που είχε πει σχετικά με την διαδικασία επιτήρηση των Πρέπει να εφαρμόζουμε μια πιο συνεπή στρατηγική τόσο για την προετοιμασία αυτών των αποστολών για την επιτήρηση των εκλογών αλλά και για την ενημέρωση που θα γίνεται κατόπιν μετά τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας πρέπει με κάθε δυνατότητα να βελτιώνουμε τον τρόπο που λειτουργούμε και να αξιοποιούμε τις πληροφορίες και τα στοιχεία που διαθέτουμε. Τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να είναι το νήμα που συνδέει όλες τις σχέσεις μας. Είναι ένας τομέας στον οποίο πρέπει να είμαστε συνεπείς. Οι κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται σε όλους με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει να αντιληφθούμε ακριβώς πώς πρέπει να γίνεται αυτή η εφαρμογή. Δεν μιλάμε για ειδικά δικαιώματα. Μιλάμε για τη δυνατότητα δυνατότητα ατόμων να έχουν, των ανθρώπων να έχουν πρόσβαση και να μπορούν να κάνουν χρήση των δικαιωμάτων τα οποία τους ανήκουν. Εκείνοι οι οποίοι σαν και εμένα έχουν εργαστεί με άτομα με ειδικέ ανάγκες γνωρίζουν πολύ καλά ότι πρέπει να ε, επιφέρουμε θετικές μεταβολές ε, σε πάρα πολλούς τομείς ώστε να μπορούν και τα άτομα με ειδικέ ανάγκες να απολαμβάνουν όλων των δικαιωμάτων που τους ανήκουν. Στην διακήρυξη για την πολιτική λογοδοσία που θα αποτελέσει στοιχείο σημαντικό της μεταρρύθμισης της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης έχω τονίσει την πρόσβαση σε στοιχεία και σε έγγραφα κάτι που θα επιτρέψει ε, στα μέλη να ενημερώνονται με πιο ολοκληρωμένο τρόπο ε, όπως έχουν ζητήσει. Δεν θέλω δομές να εφαρμοστούν δομές που θα μας ε, παρεμποδίζουν στις ε, επαφές μας με τους ε, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το, τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να είναι ένα στοιχείο οποιασδήποτε ενέργειας, οποιασδήποτε πράξης, οποιασδήποτε παρέμβασής μας. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και στη δική μας υπηρεσία. Πρέπει ε, ό, όλες οι ενέργειες, ό,τι θα κάνουμε σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα ανθρώπινα δικαιώματα να χαρακτηρίζονται από απόλυτη διαφάνεια. Η Επιτροπή είχε προτείνει αυτό που ζητήσατε. Δυστυχώς δεν εγκρίθηκε από όλα τα κράτη-μέλη. Ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προσπαθήσει να τα μεταπίσει, διότι είναι σημαντικό να συμφωνήσουν όλα τα κράτη-μέλη και ελπίζω ότι θα το θεωρήσετε αυτό σαν μια προσφορά ε, να μας βοηθήσετε για την προσχώρηση στην ε, ε, Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι κάτι που συμβαδίζει απόλυτα με την συνθήκη της Λισαβόνας και χαίρομαι που έχουμε εντολή για να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία παρόλυλα με μεμονωμένα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει. Τέλος κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ ακόμα μια φορά για την πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Σημείωσε τις σημαντικές παρατηρήσεις και παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν το έργο μου στο μέλλον και θέλω να συγχαρώ την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για ό,τι έχει ήδη κάνει. Σας ευχαριστούμε κυρία Αστόν. Κλείνουμε τη συζήτηση με την παρέμβαση της κυρίας Χαουτάλα για δύο λεπτά. Η συγγήτρια έχει το λόγο πρόεδρε. Κυρία Άστον, συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων που είναι η βάση συνεργασίας μεταξύ είπα, της εκπροσώπου και της εργασίας μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολλά και σοβαρά ελέγχθησαν Καταρχήν, για να είμαστε αξιόπιστοι, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα ίδια μέτρα και σταθμά όταν ε, αποτιμούμε τις καταστάσεις ανά τον κόσμο. Βεβαίως, ίσως υπάρχουν μικροδιαφορές και αποχρώσεις, αλλά τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν πρέπει να την χάνουν σε μεταχειρήσεις ανάλογα με τη χώρα. Επίσης πιστεύω ότι για να μπορούμε να διατρανώσουμε τη φωνή μας θα πρέπει να δούμε θέματα που μας απασχολούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν απαράδεκτες συνθήκες ε, ε, κράτηση σε φυλακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν εργαλεία βασανισμού τα οποία κυκλοφορούν Γι' αυτό πιστεύω ότι στο εγγύς μέλλον θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να ε, δούμε την συμμετοχή ορισμένων ε, κρατών μελών στις αποστολές της ΣΥΑ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Είναι πολύ λεπτό το ζήτημα, αλλά θα πρέπει να το ξαναδούμε. Ο κύριος Γκέρενς προέβαλε μια πολύ καλή ιδέα δηλαδή με την προσχώρηση στη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι 27 κυβερνήσεις θα πρέπει να δεσμευθούν να εκτελούν τις δικαστικές αποφάσεις του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτό είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για να συνεισφέρουμε Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει νέες αρμοδιότητες και θα πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε συνετά για να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να μας αποσχολήσουν εκ του σύνεγγυ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μορέιρα που συνεισφέρατε σε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστούμε κυρία Χαουτάλα. Νομίζω ότι τα χειροκρατήματα των συναδέλφων δείχνουν πόσο εκτιμούν την εργασία σας. Έχουμε λάβει έξι προτάσεις ψηφίσματα.